Άρχεται η συνεδρίαση. Άρχεται η συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι. Κολίγ Συνάδελφε Γιάτσεκ, παρακαλώ καθίστε. Ε, η κυρία Γκόμες θα ήθελε να λάβει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι παρουσίασαν οι κυρίε Ντέβα και Σιμάνσκι κάποιες τροπολογίες ε, για το θέμα των εκτρώσεων ξενοδοχείων. Ε,